Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε Ντεχούχτ. Έχει κλείσει λοιπόν η συζήτηση. Τα έξι ψηφίσματα τα οποία έχουν κατατεθεί για τη λήξη της συζήτησης από τους πράσινους, από τους, ε, τους ε, σοσιαλιστές, από τους ε, από την ΚΟΕ, από, από το ΕΛΚΑ φυσικά, από τους φιλελεύθερους και τέλος από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Αύριο στις 12 η ώρα λοιπόν θα γίνει η ψηφοφορία. Το επόμενο τώρα σημείο της διάταξης είναι η κοινή συζήτηση για τα θέματα διεθνούς εμπορίου Πρόκειται για την έκθεση Τόκια Σάφη, ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στι διεθνεί εμπορικέ συμφωνίε Α70312 κάθετο 2010. Η έκθεση Ζαντό για τι διεθνεί εμπορικέ πολιτικέ στα πλαίσια των επιτακτικών αναγκών κλιματική αλλαγή Α70310 και η έκθεση του κυρίου Ντεζίρ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στι διεθνέ εμπορικέ συμφωνίε Α70317 κάθετο 2010. Η κοινή συζήτηση λοιπόν θα ξεκινήσει από τους τρεις εισηγητές και δίνω καταρχήν το λόγο στην κυρία Σάιφη για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα αυτής της εκθέσεως συζητείται εντός της διεθνούς κοινότητας. Χώρες αναπτυσσόμενες θεωρούν ότι οι αναπτυγμένες χώρες καταφεύγουν στη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να εγκαθιδρύσουν μια μορφή προστατευτισμού αποκεκριμένου ενώ οι μένες χώρες καταδικάζουν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ των αναδειωμένων χωρών. Ήθελα να ακολουθήσουμε θετικό διάβημα, δείχνοντας πώς οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και τα εμπορικά συμφέροντα μπορούν να ενισχυθούν αμοιβαία, εάν όλες οι χώρες παίξουν σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες του παιχνιδιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει το βάρος της στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις για να επιφέρει αλλαγή θα έπρεπε να δράσει σύμφωνα με τα κείμενα των ιδιωτικών πατέρων. Σύμφωνα με αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει κυρίως στην ανάπτυξη τη βιώσιμη, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δράση της θα πρέπει, κατά την άποψή μου, ταυτόχρονα να ε, κινείται σε πολυμερή επίπεδα, διμερή επίπεδα και μονομερή επίπεδα. Στο πολυμερές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει τους διεθνείς φορείς, κυρίως την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, να λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές. Αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει παράλληλα να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ τους. Γι' αυτό προτείνω κυρίως ότι η Διεθνής, Οργάνωση, η Διεθνής Γραφείο εργασία, να έχει καθεστώς παρατηρητού εντός του ΠΟΕ. Όσον αφορά το περιβάλλον, Θεωρώ ότι η πρόσβαση στα αγαθά και την πράσινη τεχνολογία πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, διότι θα επιτρέψει όχι μόνο την πρόθεση των νέων μορφών πολιτικών όσον αφορά την απασχόληση, αλλά και νέες δυνατότητες ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είναι πολύ καλές επιδόσεις σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να εξετάσουμε το δεχόμενο δημιουργίας πραγματικής παγκόσμιας οργάνωσης περιβάλλοντος που θα μπορούσε να επεμβαίνει σε περίπτωση περιβαλλοντικού dumping σε διμερές επίπεδο, εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά μπορεί να δώσει το παράδειγμα. Χαίρομαι που συμφωνίε ε, ελευθέρων συναλλαγών νέα γενιά συμπεριλαμβάνουν ρήτρα περιοριστική τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα αυτή η πρακτική να επεκταθεί εξίσου και στο κεφάλαιο το σχετικό με την βιώσιμη ανάπτυξη. Πέραν αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται τέτοιε συμφωνίε και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει εκεί σειρά κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών που θα πρέπει να γίνονται σεβαστέ από όλου του εμπορικού εταίρους τη. Αυτέ οι βασικέ προδιαγραφέ και πρότυπα θα πρέπει να συμπληρώνονται κατά περίσταση από ε, άλλε ρήτρε ανάλογα με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική εξέλιξη τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτή η ευέλικτη και σταδιακή προσέγγιση θα επέτρεπε να αντιμετωπιστούν δικαιότερα οι διάφοροι εμπορικοί μα εταίροι και θα είναι και πιο δίκαιη προσέγγιση για όλους. Κυρίως θα πρέπει να ενισχυθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής των διμερών συμφωνιών. Προτείνω έτσι λοιπόν να γίνουν μελέτες συνεπιών εκ των προτέρων και κατά τη διάρκεια και μετά τις διαπραγματεύσεις και να μην εξετάζουν μόνο τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, ελπίζω ότι γρήγορα θα γίνουν οι εξελίξεις και στο μονομερές επίπεδο εφόσον το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων θα πρέπει πολύ σύντομα να μεταρρυθμιστεί. Όπως γνωρίζετε, επιβάλλει την κύρωση 30 περίπου συμβάσεων διεθνών για αυτό το θέμα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα για την εργασία, για το περιβάλλον και την ορθή διακυβέρνηση. Αν αυτές οι συμβάσεις επικαιρώθησαν σημαντικό βαθμό, στην πράξη δεν εφαρμόζονται καλά και επ' αυτού θα πρέπει να καταβληθούν οι προσπάθειές μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει έρευνες να καταργήσει ίσως τις προτιμήσεις ε, εάν διάφορα, διάφοροι δείχτες δείχνουν ότι οι συμβάσεις δεν εφαρμόζονται. Κλείνοντας, κάποιες από αυτές τις δράσεις μπορούν να δρομολογηθούν ήδη τώρα. Αλλά η νοοτροπία δεν θα αλλάξει σε μία μέρα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά να κινείται και σε όλα τα επίπεδα για να φτάσει σε μια πιο δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαϊφή για 4,5 λεπτά ο κύριος Λουίς Ζαντώ, Γιάννη Ζαντώ, συγγνώμη. Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σε όλους τη στιγμή ε, που μετά την συνθήκη της Λισαβόνας προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την εμπορική της πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση και να ευθυγραμμίσει με τη βιομηχανική της πολιτική το ότι ταυτόχρονα τρεις εκθέσεις ε, ε, συζητούνται στο Κοινοβούλιο για το ίδιο θέμα πολιτικό για το ίδιο πολιτικό θέμα αναρωτιόμαστε πώς το εμπόριο μπορεί να συνδεθεί με τα κοινωνικά θέματα, τα περιβαλλοντικά θέματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οποιαδήποτε συμβολή είναι ευπρόσδεκτη, διότι είμαστε σε μια ε, γενικευμένη σχιζοφρένεια. Δηλαδή, ε, στο δημόσιο διάλογο παντού ε, έχουμε με μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων, αμφισβητούνται τα κοινωνικά δικαιώματα επιδεινώνεται όλο ένα και περισσότερο το, η κατάσταση του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα ε, διαπραγματευόμαστε ε, εμπορικές συμφωνίες πολυμερείς και στον ΠΟΕ διαπραγματευόμαστε μία σειρά μέτρων που καμία σχέση δεν έχουν με τον δημόσιο διάλογο που προσπαθούν να προωθήσουν οι πολίτες. Πώς να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη στις χώρες μας σήμερα ότι ε, όταν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση παράγεται κάτι τηρώντα ε, του ε, κοινωνικού κανόνε και του περιβαλλοντικού κανόνε, μια μπάλα ποδοσφαίρου παραδείγματο χάρη και ταυτόχρονα κυκλοφορεί και στην ίδια αγορά μια μπάλα ποδοσφαίρου που έχει παραχθεί με εντελώ διαφορετικού όρου, χωρί. κανένα σεβασμό των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εντάξουμε αυτά τα κοινωνικο-περιβαλλοντικά ζητήματα στι πολυμερεί εμπορικέ συμφωνίε που διαπραγματεύονται διαπραγματευόμαστε. Σήμερα στην Ευρώπη έχουμε ε, διάφορες χώρες που λόγω των ε, εισαγωγών τους, λόγω των εισαγωγών τους λέγω, ε, αντισταθμίζουν τη μείωση των εκπομπών τους. Ε, δηλαδή ένα το 1 τρίτο των εκπομπών ε, δεν αντιστοιχούν σε παραγωγή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά οφείλονται στις αγωγές προϊόντων. Οπότε στις εμπορικές μας ανταλλαγές θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη αυτή την περιβαλλοντική διάσταση. Πώς θα εξηγήσουμε ότι θα υπογράψουμε μία συμφωνία ελευθέρου εμποδίου που θα οδηγήσει σε απερίμωση στην Κανκούνε. Τι θα κάνουμε, θα διαπραγματευτούμε μία άκαμπτη συμφωνία η οποία τελικά θα οδηγήσει σε απερίμωση στις νότιες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν όλα, να καταλάβουμε ότι είναι αλληλένδετα όλα αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδες εισηγητές όλων των πολιτικών ομάδων. Προσπαθήσαμε ε, όσο μπορούσαμε να είμαστε επικοδομητικοί. Ευελπιστώ να έχει αίσια έκβαση και η ψηφοφορία, αλλά πάντως ε, δεν είναι όλα ε, μαύρα ή άσπρα. Δεν λέμε πλέον ότι θα καταστραφούν οι βιομηχανίες επειδή προσπαθούμε να σώσουμε το περιβάλλον και επειδή υπογράφουμε αυτές τις συμφωνίες ή δεν λέμε ότι θα ασχοληθούμε μόνο με το κλίμα και θα ξεχάσουμε το εμπόριο για τον άνθρωπο άνθρακα παραδείγματο χάρη κάθε φορά προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε ε, ποιο ήταν επαπειλούμενο σε βιομηχανικό τομέα και με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να τον προστατεύσουμε. Το ίδιο ε, και στι συζητήσει που γίνονται στο ΟΜΠΟΕ για το anti-dumping επίση. Το, ε, το ίδιο έγινε με τι παραγωγικέ διαδικασίε. Για όλα αυτά τα ζητήματα από κοινού οι πολιτικέ ομάδε προσπάθησαν να καταλήξουν σε προτάσει που χάρη στι οποίε θα σημειωνόταν κάποια πρόοδο και νομίζω ότι αυτή είναι η εντολή ε, ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μόνο για όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω λοιπόν ότι αύριο αυτό το πνεύμα της επικοδομητικής ε, συνεργασίας θα οδηγήσει στην υπερψήφιση των εκθέσεων και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζουαντό. Για τέσσερα λεπτά ο κύριος Δεζίρου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω Ευχαριστώ τους συναδέρφους της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου και ιδιαίτερα τους σκιώδεις συζητητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία τους στην εκπόνηση της τρίτης αυτής εκθέσεως για να το τριών αυτών εκθέσεων μάλλον για συναφή θέματα που μας έχουν επιτρέψει να προχωρήσουμε σε σημεία που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων σε, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής. Μετά από την χρηματοοικονομική κρίση και τις συνέπειες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο υπάρχει μια συζήτηση η οποία έχει δημιουργήσει προσδοκίε των πολιτών και των πολιτικών που θέλουν να εκφράσουν τις κοινέ μα πεπιθήσει ότι στο μέλλον η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική πρέπει να οδηγήσει σε μια ρύθμιση τη παγκοσμιοποίηση και ιδίως στην επίτευξη στόχων στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Πρόκειται για κράτη και οικονομίες, αλλά κυρίως οι κύριοι φορείς σε οικονομικό επίπεδο είναι οι επιχειρήσεις. Επομένως, <clears throat> αυτό αφορά ιδιαίτερα και τις πολυεθνικές ε, επιχειρήσεις που είναι οι κύριοι παίκτε στο παγκόσμιο εμπόριο και αυτοί οι οποίοι ωφελούνται κυρίω από το άνοιγμα των αγορών. Όχι μόνο για να έχουν πρόσβαση στου καταναλωτέ, αλλά για να εξωτερικοποιήσουν ένα μεγάλο μέρο της ε, παραγωγής τους και να διαφοροποιήσουν τις πηγές τροφοδοσίας τους, κυρίως από χώρες οι οποίες δεν έχουν τις ίδιες, ε, τα ίδια πρότυπα σε επίπεδο περιβάλλοντος και κοινωνικά θέματα. Υπάρχει λοιπόν μια, ένας άγριος ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών αυτών για να προσελκύσουν επενδυτές, μια αύξηση της, του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Πολλές φορές αυτά οδηγούν σε απαράδεκτες παραβιάσεις των συνδικών εργασίας, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βλάβες στο περιβάλλον από την καταστροφή του Μποπάλ, από την Union Carbide στην Ινδία που είχε χιλιάδες θύματα. Ακόμα σήμερα υπάρχει ατιμορρησία της ε, βασικής εταιρείας. Οι, αυτά που έχουν κάνει οι εταιρείε εξόριξης πετρελαίου στη Βερμανία ή στην Αφρική που έχουν καταστρέψει το περιβάλλον και έχουν συμπεριφερθεί στους εργαζόμενους σαν σκλάβη, η εργασία των παιδιών στην κλωστοφανουργία στην ε, Ασία, η δολοφονία συνδικαλιστών στον αγροτικό τομέα στην Νότια Αμερική, όλα αυτά είναι παραδείγματα και είναι πάρα πολύ απαράδεκτα όλα αυτά γιατί οι βασικές εταιρείε είναι σε βιομηχανοποιημένες χώρες και σε αυτές περιλαμβάνονται και ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό το λόγο εδώ και πολλά χρόνια διακόπτει ο Πρόεδρος. Μήπως μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Δεν σας προφταίνουν οι διερμηνείς. Οι καμπίνες τους μάλλον δεν προφταίνουν. Λοιπόν, και επομένως από, ε, από αυτά τα προβλήματα ξεκίνησε μια συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οδηγεί στην έγκριση ψηφισμάτων από αυτή την άποψη σε ό,τι αφορά την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμή οι πρόοδοι στην κοινωνική εταιρική ευθύνη δεν έχουν οδηγήσει σε ρήτρε κοινωνικέ μέσα στι διεθνεί εμπορικέ συμφωνίε, όπω ζητάει η έκθεση ΣΑΙΦΗ. Αλλά είναι απαραίτητο διότι εφόσον υπάρχουν νομικά δεσμευτικέ ρήτρε που δεσμεύουν τα κράτη, οι εμπορικέ συμφωνίε αφορούν εθελοντικέ δεσμεύσει των επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα παράδοξο, γιατί η κοινωνική <clears throat> ευθύνη και η ευθύνη του περιβάλλοντος θα πρέπει να μα οδηγήσουν σε μια παγκοσμιοποίηση η οποία σέβεται περισσότερο την αηφόρο ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Θέλουμε λοιπόν αυτή η εταιρική ευθύνη να ενσωματωθεί στι συμφωνίε εμπορίου και να υπάρξει συγκεκριμένα μια ρήτρα κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων μέσα στο κεφάλαιο τη αηφόρου ανάπτυξη, ιδίω για τι αναπτυσσόμενε χώρε που να είναι σαφή και επαληθεύσιμη δέσμευση των επιχειρήσεων. υπάρχει μια αμφίδρομη δέσμευση λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των επιχειρήσεων για να μπορέσουν οι επιχειρήσει αυτέ να αναλάβουν ε, υποχρεώσει οι οποίε θα είναι επαληθεύσιμε. Να υπάρχουν σημεία επαφή για να μπορούν να δίνονται πληροφορίε, αλλά επίση να λαμβάνουν υπόψη και οι μαρτυρίε τη κοινωνία των πολιτών, των συνδικαλιστών να υπάρχει μια υποχρέωση να δίδεται ένας απολογισμός για όλα αυτά και να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει επίσης και η εύλογη φροντίδα από τις πλευρά των επιχειρήσεων για να προλαμβάνουν τέτοιες παραβιάσεις και ιδίως να μπορούν να αποφευθούν παραβιάσεις της, κοινωνικής, της ε, κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων αλλά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βλαβών προς το περιβάλλον. Πάλι ο πρόεδρος διακόπτει. Σας ευχαριστώ κύριε Ντεζίρ. Ζητώ την επίγειά σας, αλλά ορισμένα πράγματα δεν γίνονται. Έχετε τέσσερα λεφτά, έχετε ξεπεράσει τα μισή. Και παρά το γεγονός ότι σας διέκοψα, προσπαθώ να είμαι δίκαιος με όλους τους βουλευτές, αλλά έχετε, έχετε <laughs> υπόψη σας ότι δεν σημαίνει το να φροντίζει κανείς τον χρόνο του να διαβάζει πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να προλάβει κανείς να καταλάβει. Αυτό δεν αφορά μόνο τα γαλλικά, άφερα όλες τις ομιλίες διότι περνάνε από τις καμπίνες, από του διερμηνείς. Και αν δεν μπορούν οι διερμηνείς να προλάβουν, τότε οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά που λέτε, ακριβώς γιατί διαβάζετε πάρα πολύ γρήγορα την ομιλία σας. Σας παρακαλώ λοιπόν να περιοριστείτε στο χρόνο αγόρευσή σας και να μην περιορίζει το χρόνο σκατσουδιάς στη συνέχεια. Διαδικαστική παρέμβαση. Πρόεδρε, είναι η δεύτερη φορά που είμαι σε αυτή την αίθουσα και είδα τον Πρόεδρο να διακόπτει έναν από τους αγορητές επί τη βάση της ταχύτητας της αγορεύσεως. Δεν ξέρω πώς συχνά μιλάτε εσείς ο ίδιος. Πρέπει να καταλάβετε όμως αυτή η διακοπή έχει τη συνέπεια να καταστρέφει την ομιλία. Διαφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει ο κύριος Ντεζίρ, που είπε ο κύριος Ντεζίρ. Αλλά οι διερμηνείς πληρώνονται, είναι πληρωνόμενοι εργαζόμενοι και αν δεν μπορούν να προλάβουν δικό τους το πρόβλημα και δεν πρέπει ο πρόεδρος να διακόπτει όπως διακόψατε εσείς πριν. Αυτό είναι το καθήκον μου αγαπητέ συνάδελφε, λέει ο πρόεδρος. Εμείς πληρώνουμε εκατομμύρια για να κάνουμε αυτά που κάνουμε σε, αν σε 10 λεπτά μπορούμε να πούμε κάτι που κοστίζει ένα εκατομμύριο, δεν μπορούμε να το κάνουμε με 100 εκατομμύρια σε 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, εγώ ε, γνωρίζω πολύ καλά, γιατί υπήρξα βουλευτή, γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχει ένα σημείο πέραν του οποίου οι βουλευτές δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και οι βουλευτές χρησιμοποιούν την δυνατότητα που υπάρχει να ζητήσουν από τον Πρόεδρο να, να ζητήσει από τον ομιλητή να μιλάει πιο, ε, πιο αργά. Εάν λοιπόν δεν μπορεί να μεταφραστεί μια ομιλία, αυτό έχει επιπτώσει σε όλους. Κυρία Μπερές. Επιτρέπω στον εαυτό μου αυτό το οποίο επιτρέπετε και εσείς στη δική σας επιτροπή, δηλαδή να αντιμετωπίσω θέματα που είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως γίνεται σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή γίνεται και στην, στην Ολομέλεια. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντεχούχτ. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σε διαβεβαιώνω ότι αν ποτέ θα έτρεχα τα 100 μέτρα θα, μου, θα χρειαζόμουν τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους εισηγητές και την Επιτροπή Ίντα για τις εκθέσεις. Θέτουν σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τη βολή της εμπορικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς την επίτευξη κάποιων από τους θεμελώδεις στόχους ε, της δημόσιας πολιτικής, το σεβασμό των θρύπων δικαιωμάτων, την επιδίωξη οικονομικής ευμάρειας και κοινωνικής δικαιοσύνης, την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, το σεβασμό του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του κλιματολογικού συστήματος θα πρέπει να καταλάβετε ότι το σύντομο χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μου σήμερα είναι αδύνατο να επισέθω σε λεπτομέρειε κάθε θέματο. Αλλά επιτρέψτε μου να προβώ σε κάποιε γενικέ ε, δηλώσει. Οι τρει εκθέσει έχουν πολλά κοινά σημεία. Όλε ασχολούνται με τη συνοχή των πολιτικών και αναφέρονται στην ανάγκη η εμπορική πολιτική να διεξάγεται στα πλαίσια των γενικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ιδιαίτερα οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών τέτοιων στόχων. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω παραπάνω με το στόχο να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να πετύχουμε τους εν λόγω στόχους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τονιστεί ότι η αποτελεσματική δράση θα πρέπει να βασίζεται επί των μέσων εκείνων που είναι τα πλέον ε, ικανά να πετύχουν τους στόχους. Η εμπορική πολιτική είναι βασικό φορέα που μπορεί να προωθήσει το κοινωνικό μοντέλο και να το διαφυλάξει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, τι αξίε και τι αρχέ αυτού. Και ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλε προσδοκίε σχετικά με αυτό το θέμα θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να επιληθούν απαραίτητα μέσω τη εμπορική πολιτική και άλλε πολιτικέ που να προσφέρουν καλύτερε δυνατότητε για αποτελεσματικέ λύσει. Θα πρέπει επίση να γνωρίζουμε ότι η εξισορρόπηση διαφόρων συμφερόντων είναι στο επίκεντρο τη πολιτική δράση και πάντα θα υπάρχουν επιλογέ που θα πρέπει να γίνουν. Προκλήσει επίση θα διαφέρουν. Ανάλογα με το κατά πόσο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόνομα μέσα όπως είναι τα συστήματα γενικών προτιμήσεων, γενικών προτιμήσεων, πολυμερείς ή μονομερείς ε, προ, ε, διμερείς συμφωνίες. Η αναφορά της κυρία Σαΐφη για τα κοινωνικά δικαιώματα σε εμπορικές συμφωνίες αναγνωρίζει ότι όλες αυτές οι διαστάσεις που παρέθεσα προσφέρουν διαφορετικές δυνατότητες. Εν γέννη, η διεθνή συνεργασία έχει τη δυνατότητα να προωθήσει πιο αποτελεσματικέ δράσει. Από την άλλη πλευρά, πρέπει, χρειάζονται δύο άνθρωποι για να χορέψουν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τι είναι αποδεκτό για να, να βρούμε τέρους και σε πιο με ποιο τίμημα, κυρίως όσον αφορά τις πολυμερείς διευθετήσεις. Η επίτευξη της συνένεσης εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βελτιώσει τη διεθνή διακυβέρνηση, τη συμφέρει αυτό, και μέσω αυξημένη συνοχής μεταξύ δράσεων σε διάφορα βήματα. Στα φόρα, στο ΠΟΕ, στο Διεθνέ Γραφείο Εργασίες, στο Φορέα για τις συζητήσεις της Διεθνής για το κλίμα, οι τρεις εκθέσεις σκιαγραφούν τρεις διαφορετικούς τομείς θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να μπορέσουμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ των πρακτικών βηγμάτων που μπορούν να είναι επιτυχή βράχη πρόθεσμα και εκείνων που πλέον μακροπρόθεσμα θα πετύχουν τους στόχους τους. Θα πρέπει να μας δώσουμε περιθώριο για να σκεφτούμε στο μέλλον. Θέλουμε αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω πολιτικής. Το ίδιο ισχύει και στις διμερείς συμφωνίες. Οι διατάξεις της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου δεν είναι απλώς δηλώσεις καλών προθέσεων, πρέπει να εφαρμόζονται, να είναι εφαρμόσιμες. Στρεφόμενο προ τον κύριο έκθεση του κυρίου Ζαντό για την αλλαγή του κλίματο, να αναφέρω την ανάγκη που υπάρχει να εξασφαλίσουμε ότι εσδήποτε επιλογέ πράγματι θα μπορέσουν αποτελεσματικά να μειώσουν τον κίνδυνο διαρροή διοξιδίου του άνθρακο και να μπορούν με λογικό κόστο να εφαρμόζονται. Όλοι γνωρίζουμε, παραδείγματο χάρη, ότι επιλογέ όπω τα μεθοριακά ε, μέτρα δημιουργούν διάφορα ζητήματα. Πώ να προσμετρήσουμε, να παρακολουθήσουμε κλπ ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να αξιολογήσουμε όλα τα θέματα πριν να θέλουμε να προχωρήσουμε βιαστικά σε συμπεράσματα. Τούτων λεχθέντων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να εξετάζει όλες τις εφικτές λύσεις. Όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Ντεζίρ περί της κοινωνικής ευθύνης των εταιριών είπε ότι οι πρωτοβουλίες τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να υποστηρίζουν παρά να ρυθμίζουν τι δραστηριότητε αυτέ. Όμως υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ υποστήριξης, ρύθμισης και επιβολής. Μια γραμμή την οποία ο με επιδεξιότητα την εξέταση, αλλά συνεπάγεται διάφορες πτυχέ που θα εξεταστούν, κυρίω την πολιτική. Το CSR δεν μπορεί να εξαιρεί χώρε από τις ευθύνε που έχουν ε, ε, όσον αφορά την επιβολή των νόμων του. Όπω και οι κρατικοί φορεί δεν είναι εκεί να επιβάλλουν την εταιρική πολιτική αυτή καθ' αυτή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλά από αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στην επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του ΩΣΑ όσον αφορά τι πολυεθνικές επιχειρήσει κάτι που πρέπει να υιοθετηθεί κανονικά το 2011. Αυτό είναι ένα παράδειγμα τη χρήσιμου έργου που επιτελείται και στο οποίο συμμετέχουμε ενεργά. Οι εκθέσει που συζητούνται σήμερα συμπεριλαμβάνουν πολύ συγκεκριμένου προσανατολισμού, όσον αφορά διόδου που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να βελτιώσουμε αποτελεσματικότητα, τη συνέπεια, το πεδίο εφαρμογή και τη διαφάνεια των δράσεών μα όσον αφορά κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα στι διάφορε συμφωνίε και διατάξει για το CSR και για τα θέματα αλλαγή του κλίματο. Βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάζει αυτέ τι πτυχέ συνεχώ και θα εξετάσει και του προσανατολισμού που σκιαγραφούνται. Υπό του όρου που προανέφερα, θα πρέπει να περιμένετε ότι θα έχουμε αρκετέ επιφυλάξει σε σημαντικά σημεία και θα συμφωνούμε και απόλυτα βέβαια σε άλλα σημεία των εκθέσεων. Θα υπάρχει κάθε δυνατότητα στα πλαίσια τη αναθεωρήσεω του συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων του χρόνου να συζητήσουμε του επόμενου μήνε και έτη τα θέματα αυτά περαιτέρω. Και στα πλαίσια των επικειμένων ε, διαδικασιών των νομοθετικών τη Συμφώνου Γνώμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να εξετάσει μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σωστά μέσα, αποτελεσματικά μέσα, εφαρμόσιμα μέσα, ούτω ώστε η εμπορική μας πολιτική να αντικατοπτρίζει διάφορε κοινωνικές ανησυχίε. Βασική αρχή θα πρέπει να είναι προσεκτική αναλυτική διαμόρφωση πολιτικής επί τη βάση ε, ε μελλοντικής αναλύσεως και ρεαλιστικών προσδοκιών. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ακολουθούν οι ομιλητέ εξ των Επιτροπών, ο κ. Μάρτιν από την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου για δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, εάν θέλει, θα πρέπει να, επιτυχά, να επιτύχει το μέγιστο δυνατό κέρδο ή θα πρέπει να επιτύχει στόχου όπω είναι το, η αηφόρο ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά πρότυπα και δημοκρατικέ αρχέ οι τρεις ομιλητές πριν από μένα είπαν ότι είναι το δεύτερο το οποίο πρέπει να προέχει και το τόνισε και η Κομισιόν. Ήδη στις δράσεις μας εμείς θέτουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τα εργασιακά πρότυπα σαν στοιχεία των διμερών συμφωνιών μας. Το ερώτημα είναι το πράττουμε αυτό όμως με έναν τρόπο ο οποίος μα επιτρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά και θα υπάρχει συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει μεγάλε αμφιβολίε για το πόσο ευσταθεί κάτι τέτοιο. Θα θέλαμε στο μέλλον σε μελλοντικέ εμπορικέ συμφωνίε να εξασφαλίσουμε ότι πρωτού μονογραφηθεί η οποιαδήποτε συμφωνία θα γίνει μια ε, έρευνα αντικτύπου για να ξέρουμε ότι όχι μόνο θα προκύψουν ε, εμπορικά και οικονομικά ωφέλη, αλλά και ωφέλη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το σύστημα για την αναστολή συμφωνιών λόγω παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνει πιο προσπελάσιμο και αξιόπιστο και εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι ο κύριος Ντεχούχτε έχει ακολουθήσει αυτή την οδό στην συμφωνία με την Κορέα. Επίσης, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ θα πρέπει να υπάρχει μια πιο δίκαια βαθμονόμηση των ε, εταίρων μας ώστε η εφαρμογή των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ε, αναπτυξιακών στόχων θα επιτυγχάνει. Η κυρία Σάιφη, ο κύριος Ζαντό και ο κύριος Ντεζίρ τόνισαν ότι δεν είναι αυτός σκοπός το εμπόριο, ότι πρέπει να είναι αντίθετα τμήμα μιας ευρύτερης πληρέστερης στρατηγικής για να προωθήσουμε ένα πιο ισοδίκαιο, υγιέστερο και πιο ειρηνικό πλανήτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μάρτιν. Για την Επιτροπή Ανάπτυξη έχουμε δύο μιλητές, καταρχήν ο κ. Κατσμαρέκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που ο Επίτροπος Ντεγκούχτ, καθώς και οι συγγητές των τριών εκθέσεων, κατανοούν ότι ε, για να ε, κατοχυρώσουμε κοινωνικά περιβαλλοντικά πρότυπα θα πρέπει να ε, προωθήσουμε τα πρότυπά μας ε, ε, όχι μόνο στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου αλλά και στα πλαίσια της αναπτυξιακής ε, συνεργασίας. Έχουμε υποβάλει κάποια σχόλια για την έκθεση ΣΑΙΦΗ ε, ως προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχουν κάποιες χώρες που παραμελούν ε, το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά πρέπει επίσης να σεβόμαστε και τους, τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Αν μου επιτρέπετε, εξ ονόματο τη Επιτροπή Ανάπτυξη, θα ήθελα να δώσω ορισμένε από τι κατευθυντήρε γραμμέ στην Επιτροπή μα, να τονίσω ότι για την κλιματική αλλαγή η πιο φτωχέ χώρε είναι αυτέ οι οποίε είναι και οι πιο ευάλωτε. Η συμμετοχή του λοιπόν στην εκπώνηση πολιτικών, ιδίω εμπορικών πολιτικών, είναι ουσιώδης. Θέλω να τονίσω επίση ότι η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι αφορά το εμπορικό τα εμπορικά θέματα πρέπει να συνάδει με τον αγώνα εναντίον τη κλιματική αλλαγή και τη ένδυας. Πρέπει μέσα να υπάρχουν ρήτρε για το περιβάλλον σε όλε τι εμπορικέ συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρξει αναθεώρηση των μηχανισμών καθαρή ανάπτυξη, ένα πραγματικό μηχανισμός μεταλαμβάνευση της ε, τεχνολογίας και αγώνας κατά της πειρατείας. 20% των μεταφορών που από τις μεταφορές θα πρέπει να μειώσουμε τις μετακινήσεις προϊόντων, ιδίως στη γεωργία, για να μπορέσει να υπάρχει τοπική <clears throat> απασχόληση και για μας και τις αναπτυσσόμενες χώρες και μείωση των εκπομπών του Θεμοκηπίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέζ για την Επιτροπή Απασχόλησης, η κυρία Μπερέσ. Πρόεδρε, επί, Επίτροπε, ε, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης, ε, θα συμφωνήσουμε με την έκθεση Ντεσίρ από την Επιτροπή Ίντα και στην Επιτροπή μας ε, όπως και σε άλλες, το πιο πολύ συζητημένο θέμα είναι σε τι ωφελεί η εταιρική ευθύνη. Είναι αυτοσκοπός ή θα πρέπει να οδηγήσει σε νομοθετήματα εφόσον εφαρμόζεται από πολλές επιχειρήσεις. Ακόμη δεν έχει απαντηθεί αυτό το θέμα και θα πρέπει να το δούμε στο γενικότερο πλαίσιο της διακυβέρνησης των εταιριών. Στην Επιτροπή Απασχόλησης θεωρούμε ότι αυτή η κοινωνική εταιρική ευθύνη είναι ε, κέρια σημασία εάν θέλουμε στα πλαίσια των πολυμερών συμφωνιών ε, να καταπολεμήσουμε την παράνομη εργασία ή τη φοροδιαφυγή. Θα πρέπει επίσης ε, για να αξιοποιήσουμε και να προαγάγουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη, να φροντίσουμε ώστε τα συμβούλια εργαζομένων ε, στις εταιρείες και η διοίκηση των εταιρεών να κινητοποιηθούν. Τα επιχειρησιακά αυτά συμβούλια έχουν αποφασιστική συμβολή ε, για να ε, μην ξεχνάμε επίσης ε, και ότι στον ΟΗΕ αναγνωρίζεται ο βασικός ρόλος αυτής της εταιρικής κοινωνικής ε, ευθύνης. Πιστεύουμε πως αυτή η εταιρική ευθύνη είναι και ένα εργαλείο ανταγωνιστικότητας και οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε παρότι καταλήγουμε σε συνένεση μόνο όταν ε, προσδιορίζουμε αυτή την ευθύνη βασισμένη σε κοινώ αποδεκτά πρότυπα. Δεν μπορούμε δε να αντικαταστήσουμε ε, τις συλλογικέ συμβάσεις ε, με πρόσχημα αυτή την κοινωνική ευθύνη. Τέλος, αυτή η κοινωνική ευθύνη ακόμη και στις εμπορικές συμφωνίες πρέπει να είναι δυναμική και να προσαρμόζεται όταν πρέπει να καλύψουμε και άλλους τομείς. Ευχαριστούμε κυρία Μπερές. Δυόμιση λεπτά από την Κοινωνική Επιτροπή. Κύριος Άουιτς σαν εισηγητή του Κοινοβουλίου για την, εταιρική την κοινωνική ευθύνη των εταίρων, επί τρει θητείε κοινοβουλευτικέ, καλωσορίζω την πρωτοβουλία του κ. Ντεζίρ για το εμπόριο και το CSR. Οι εταιρείε πολύ συχνά λένε ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουν αυτή την τυχή στη πολιτική του και αυτή η πρωτοβουλία ε, δείχνει ότι και η δημόσια πολιτική πρέπει να το ίδιο και ελπίζω και ο Επίτροπο κ. Ντεχούκτ ε, που ε, έκανε κάποιες συστάσεις, αν το λάβει αυτό υπόψη Τα πρόσφατα χρόνια η δουλειά μου όλο και περισσότερο αφορούσε την εκπροσώπηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων στην πρόθεση παγκοσμίων συμφωνιών και μηχανισμών CSR. Γι' αυτό σαν φρένο του καθεντηρίου γραμμών του ΟΣΑ είναι το καλύτερο πρότυπο των CSR και κάτι που έχουν προσυπογράψει οι κυβερνήσει. Και γι' αυτό υποστηρίζω την παράγραφο 25 για τη μελλοντική εμπορική συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ενώσης που θα πρέπει να, υπογρά... να ακολουθεί αυτέ τι κατά γραμμέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσημα σημεία επαφή όσον αφορά ε, αυτό το θέμα στα πλαίσια αυτών των προδιαγραφών. Ήμουν σύμβουλο του καθηγητού Τζον Ράικεϊ όσον αφορά τι επιχειρήσει και ανθρώπινα δικαιώματα και εγκρίνω την απέτηση που αναφέρεται στην έκθεση εταιρείε να αναλάβουν ε, υπόψη στην ιδιωτική σκέψη Q αυτού του θέματο. Οικοσορίζω την, την υποστήριξη τη Σουηδική ε, Προεδρία για τι συστάσει τη ΥΠΑ τη εκπροσώπου που συμπεριλαμβάνεται στη συμπεράσματα του Συμβουλίου. Επίτροπο θα πρέπει ιδιαίτερω να διαβάσει τι επικρίσει των κυβερνητικών αποτυχιών όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στις, όσον αφορά τι επενδύσει και σαν μέλος του Συμβουλευτικού Φορέα για την Πρωτοβουλία καλά να φέρει στην παράγραφο 15 διαφάνεια, αλλά επίση θα ήθελα να ζωτήσω ότι η δημόσια διαβούλευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πήγε τη αφορά την μία αποκάλυψη των οικονομικών στοιχείων να ε, ακολουθεί την, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα το θέμα του σεβασμού του απορρίτου των διαφόρων πληροφοριών που χορηγούνται για να προωθηθούν αυτέ οι πολιτικέ. Σα έχω πει ότι μερικές φορές αναγκάζομαι να διακόψω συναδέλφο. όταν μου λένε οι διερμηνεί όμω ότι μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Σα παρακαλώ να μιλάτε με φυσιολογικό ρυθμό ομιλίε. Ακολουθεί ο κ. Κασπάρη από την ομάδα του ΕΛΚ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Βίλαντ, αγαπητοί συνάδελφοι, Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τους τρεις συγητέ για τις εκθέσεις τους. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή και η κοινή συζήτηση των τριών αυτών εκθέσεων είναι πολύ καλό παράδειγμα της θέσης του Κοινοβουλίου για αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Θέλω να εστιάσω την προσοχή μου σε ένα σημείο. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτά τα τρία, σε αυτές τις τρεις εκθέσεις αντιμετωπίζουμε το πώ η εμπορική πολιτική μπορεί να συμβάλλει στου τρει αυτού τομείς που, αναβάλαμε, που αναφέραμε περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και κοινωνική ευθύνη. Η κυρία Σάιφη αναφέρθηκε στα ανθρώπινα δικαιώματα, ο κύριο Ζαντό στα κλιματικά θέματα και ο κύριο Δεζή στην κοινωνική ευθύνη. Όλα αυτά τονίζουν λοιπόν το ρόλο που μπορεί να έχει το εμπόριο για όλα αυτά τα θέματα. Αλλά θα ήθελα επίση να κοιτάξουμε και τι κάνουν και οι πολιτικές αυτές οι πολιτικές περιβάλλοντος, η πολιτική κλιματικής αλλαγής, η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνουν υπόψη τους και την εμπορική πολιτική. Υπάρχει μια ενιαία στα ε, στοχοθεσία. Γιατί δεν γίνεται πολλές φορές και μια προσπάθεια να κατανοήσουν και το ρόλο της εμπορικής πολιτικής. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει ότι παραδείγματο στην Κοπεχάγη δεν καταφέραμε να επιτύχουμε μια ε, λύση στα κλιματικά θέματα. Δεν μπορούμε να υπερφορτώνουμε λοιπόν την εμπορική πολιτική με την επίλυση προβλημάτων τα οποία δεν έχουν καταφέρει αυτόνομα να λύσουν όλε αυτέ οι επιμέρου πολιτικέ. Ελπίζω λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει στου επόμενου μήνε να τονίσει και το ρόλο που πρέπει να έχουν οι επιμέρου αυτέ πολιτικέ και για την υποστήριξη τη εμπορική πολιτική. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε και την αντιμετώπιση των εμπορικών θεμάτων και όχι να συζητάμε όλα τα άλλα εκτό από το εμπόριο. Ευχαριστώ κύριε Κασπάρη. Για τους σοσιαλιστές, ο κύριος Άσενς, για ένα, Ασένς, για ένα λεπτό. Πραγματικά πολλές φορές ε, είμαι σίγουρος ότι οι υπηρεσίες σας θα σας εξηγούν πώς δεν είναι δυνατόν να ληφθούν και να εφαρμοστούν κάποια μέτρα που είναι απαραίτητα για την κλιματική αλλαγή. Όμως η απειλή της κλιματικής αλλαγής είναι τόσο τεράστια ε, που δεν είναι το θέμα ε, πώς, ε, τι θα εφαρμοστεί, αλλά το θέμα είναι πώ θα βρούμε του τρόπου για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, πώ θα βρούμε του τρόπου να εφαρμόσουμε τα απαραίτητα πράγματα. Μια ε, λύση που συζητιέται είναι και όσον αφορά την συμβολή του εμπορίου στην κλιματική αλλαγή είναι τα border tax adjustments. Με λίγα λόγια, τη φορολογία επί ε, εισαγωγών ε, από χώρε που δεν παίρνουν τα μέτρα με εμά αναφορικά με την κλιματική αλλαγή. Επίση, θα πρέπει να εξετάσουμε αντικίνητρα για την εμπορία ομοειδών ειδών το νερό είναι ένα τοπικό σπόρο και όμω χώρε όπω παραδείγματο χάρη η Γαλλία ή το Βέλγιο είναι την ίδια στιγμή από του μεγαλύτερου Ευρωπαίου εξαγωγέ και του μεγαλύτερου Ευρωπαίου εισαγωγεί νερού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί για δύο μισή λεπτά από την ομάδα των Φιλελευθέρων και, Μετα... και Δημοκρατών ο κύριος Καζάκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές ΣΑΕΦ, Ντεζίρ και Ζαντό. Ε, ήταν εξαιρετική η εργασία που έκανα και για τις τρεις εκθέσεις. Καλωσορίζω την ιδέα βάση της οποίας ε, δεσμευτικές ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και θα πρέπει να μεριμνούμε ώστε να εφαρμόζονται σωστά αυτές οι ρήτρες. Ε, κυρίως για τα εργασιακά δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών θα ήθελα να σας μιλήσω στα πλαίσια της σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, το απλό και το ΣΥΝ, ε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προαγωγή των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να υπάρχει άμεση σύνδεση ε, σε αυτές τις συμφωνίες ανάμεσα στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ και τις Ερήτρες προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίσης ανάμεσα στον ΟΗΕ και το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και τον ΠΟΕ θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία και θα πρέπει να έχει καθεστώς παρατηρητού στα πλαίσια του Κατά τη γνώμη μου επίσης, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται αρκούντος για τις προϊούσες διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να ασκήσουμε τις νέες εξουσίες που προσέδωσε η συνθήκη της Λισαβόνα στο Κοινοβούλιο. Για την έκθεση του κυρίου Ζαντό, φυσικά θα πρέπει να Επραγάγουμε το πράσινο εμπόριο, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε πώς ακριβώς χαρακτηρίζουμε κάποιο προϊόν ως πράσινο ε, και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και για τις ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειες. για την τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων. Επίσης θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυξάνει ε, το κόστος της παραγωγής. Ε, δεν προβλέπεται ε, να επιτευχθεί συμφωνία για κατά των κλιματικών αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί ήδη από μόνη της, να έχουμε δεσμευτικούς ε, στόχους Κλείνοντας θα ευχαριστήσω και τους τρεις εισηγητές ε, και ελπίζω ότι θα επηρεαστούν ε, οι ε, διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Σας ευχαριστούμε κύριε Κάζακ. από πλευράς των Πρασίνων, ο συνάδελφος Τέιλορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και συνάδελφοι. Ήμουν ο Σκιώδης των Πρασίνων και την έκθεση Σαΐφη και την έκθεση Ντεζίρ. Ευπρόσδεκτε και δύο είναι σημαντικά βήματα πρόοδου. Θα εξασφαλίσουμε καλύτερα ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικέ και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και πρότυπα στις χώρες ε, που είναι τέρη μα εμπορική. Αν αυτές οι χώρες θέλουν να πουλήσουν στην ε, κερδοφόρα ε, αγορά τη Ευρωπαϊκή τα θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν αξιοπρεπεί και βιώσιμε προδιαγραφέ στι στις του και να εξασφαλίσουμε μέσω υποχρεωτικών ρητρών και απαιτήσεων βελτιώσει. Αυτέ θα συμπεριλαμβάνονται στι εμπορικέ συμφωνίε. Αυτό είναι ένα τρόπο να το πετύχουμε αυτό. Ο κ. Σάφη έκανε πολύ καλή δουλειά σαν εισηγήτρια και συζητεί τα διάφορα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων σε διαφορετικά επίπεδα. Συμφωνήσαμε λοιπόν με τις προτάσεις ΣΑΦΗ ότι ένας παγκόσμιος οργανισμός περιβάλλοντος θα πρέπει να δημιουργηθεί και διεθνώ Γραφείο εργασία θα πρέπει να ενισχυθεί, να αυξηθεί το, η θέση που έχει. Και το κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη στα FDA είναι κάτι πρόσδεκτο, αλλά αυτά τα πρότυπα θα πρέπει να είναι δεσμευτικά και όχι εθελοντικά. Και τα συστήματα γενικευμένων προτιμήσεων θα πρέπει να έχουν πράγματι δύναμη και να μπορούν να εφαρμόζονται. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όμως με τον συγκητή ότι η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο FTI με την ε, Κολομβία ήταν ικανοποιητικό. Ε, εγώ νομίζω ότι ήταν απλώς ε, μια τυπική ρήτρα που γελιοποιεί τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό το θέμα. Τώρα στρεφόμενος προς την έκθεση του κυρίου Ντεζίρ, πρέπει να πω ότι δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο με αυτά που λέει όταν κατονομάζει τις ε, διεθνείς επιχειρήσεις ως πηγή αρνητικών συνεπειών όσον αφορά το περιβάλλον και τα κοινωνικά μας πρότυπα. Έχουν κερδίσει πολλά από την απελευθέρωση του εμπορίου, έχουν εκμεταλλευτεί τα φθηνά εργατικά χέρια και πολύ συχνά τα φθηνά υλικά. Αλλά δεν αναδιανέμουν με επαρκή τρόπο τον πλούτο που δημιούργησαν εις βάρος των άλλων. Τροποποίησαμε επιτυχώ και τι δύο εκθέσει και θα υποστηρίξουμε και τι δύο όσον αφορά την ψηφοφορία. Κλείνοντα, εντάχει να τονίσω ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι κοινωνικές ευθύνες ε, να λάβουν προτεραιότητα και να βάλουμε ποια θέματα έχουν προτεραιότητα για μα μέσω υποχρεωτικών απαιτήσεων και να μην βασιζόμαστε επί που χρησιμοποιούνται θελοντικά. Merci κύριε Τέιλορ για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές ο κ. Βαντάλεν για 1,5 λεπτό. Είναι πολύ καλή η έκθεση ε, Ζαΐφη. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και στο μέλλον με τις σχέσεις με άλλες χώρες και οι συμφωνίες με άλλες χώρες δεν θα πρέπει να γίνονται ε, ει βάρο των κοινωνικών προδιαγραφών. Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι κοινωνικέ ρήτρε. Έχει σχέσει οικονομικέ με το Πακιστάν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν αυτή η χώρα ε, να έχει οικονομικά ωφέλη από αυτή τη σχέση για να μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και μέσα από πλημμύρε. Χρειάζεται λοιπόν όμως να ατροποποιηθεί να έχει σωστή νομοθεσία, όπως είναι για την βλασφήμια, παραδείγματο χάρη. Είναι αναχρονιστικά τα μέτρα. Και θα πρέπει λοιπόν να μην δεχόμαστε μέτρα τα οποία δεν έχουν ε, σχέση με τις εμπορικές σχέσεις. Λοιπόν, θα πρέπει οι επενδύσει και τα εμπορικά συμφέροντα να ε, λαμβάνονται υπόψη μαζί με τι κοινωνικέ προδιαγραφέ. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι είχαμε πει και στο ψήφισμά μα του Μαρτίου 2010. Ευχαριστώ, κ. Βαντάλεν. Επόμενο για δύο λεπτά. Για την ΚΟΕ. Ο κ. Σόλτ μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Ντεχούχτ, έντιμοι συνάδελφοι, οι τρεις αυτές ε, ε, εκθέσεις δεν είναι τυχαία σε μια κοινή συζήτηση και θέλω καταρχήν να συγχαρώ τους τρεις ε, εισηγητές. Όλοι τονίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ανεξάρτητα από πολιτικές ομάδες θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά με ένα κοινό τρόπο αντιμετώπισης. Έχουμε σημαντικές προκλήσεις ε, ενώπιόν μας και γι' αυτό είναι μια πάρα πολύ επίκαιρη και εύστοχη συζήτηση γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται το θέμα της εμπορικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια ευκαιρία για να έχουμε πολλές σκέψεις και πολλές συγκεκριμένε προτάσεις για σχέδια και προγράμματα. Προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπερπίδηση της, ε, υπερκέραση της ένδυας, αυτά είναι σημαντικά καθήκοντα για όλους μας. Αυτά είναι πιο σημαντικά από τα εμπορικά συμφέροντα. Πρέπει η σύγχρονη εμπορική πολιτική να ενσωματώσει όλες αυτές τις βασικές ιδέες να εξασφαλίσουμε την ευμάρεια με την έννοια του Human Development Index της ανθρώπινης ανάπτυξης και να εξασφαλίσουμε και το κράτο δικαίου. Και μόνο έτσι μπορεί να είναι επιτυχής και η ευρωπαϊκή οικονομία και να μπορεί να διαδικτυωθεί με άλλες οικονομίες όλου του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα εμπορικός ανταγωνισμός η ομάδα μου θα ήθελε να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο οι εισηγητέ. Παραδείγματο χάρη, αναρωτιέμαι αν είναι αρκετό οι επιχειρήσεις μόνες τους εθελοντικά να θεσπίζουν την ε, δική τους ε, εταιρική ευθύνη όταν εκατομμύρια άτομα όλου του κόσμου εξαρτώνται από αυτόν. Όταν υπάρχει εκμετάλλευση ε, πόρων, όταν υπάρχει εκμετάλλευση παιδικής εργασίας, όταν προϊόντα καθημερινά όπως η σοκολάτα παράγονται σε σκανδαλώδες συνθήκες. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη τροφοδοσία με πρώτες ύλες, όπως είπατε κύριε Επίτροπε, αυτό απαιτεί να λάβουμε υπόψη και τις πτυχές των τριών αυτών εκθέσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Για ένα λεπτό για την ομάδα Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ο Earl of Dartmouth. Κύριε Πρόεδρε, το εμπόριο δίνει αμοιβαία ευμάρια και τονίζω το αμοιβαίο. <clears throat> Ω εκ τούτου η εμπορική πολιτική σχεδόν ποτέ δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται με πολιτικέ ατζέντε. Προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ του τρει εισηγητέ αλλά η φιλοσοφία που διατρέχει αυτές τις εκθέσεις έχει παρουσιαστεί σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και έχει καταψηφιστεί τις περισσότερες φορές. Εδώ βλέπουμε μια προσπάθεια χειραγώγησης της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δυστυχώς δεσμεύει και το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή για να μπορέσει λαθρέως και λάθραν να περάσει μια κοινωνική ατζέντα η οποία έχει απορριφθεί σε πολιτικό επίπεδο. Οι μηχανογραφίες των εισηγητών είναι εντυπωσιακέ. Αλλά ως δημοκράτης πρέπει να πω όχι και γι' αυτό θα πούμε όχι σε αυτές τις εκθέσει αύριο. Σας ευχαριστώ κύριε Έρλα για τους μη εγγεγραμμένους η κυρία Στάσεν για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε οι αιτίες και οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών βασίζονται σε μια επιστημονική θεωρία, αλλά τελικά έχει γίνει ηθολογικό το ζήτημα, θρησκευτικό. Στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου μιλάμε για την κλιματολογική διπλωματία. Ε, θέλει να διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέτρο όμως ε, που ε, ικανοποιείται από όλε τι διατάξεις των προτινόμενων σχεδίων. Οι χώρες θέλουν να εξαγάγουν, άλλες θέλουν να εισαγάγουν. Ξέρουμε οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα κατά πόσο πλήττουν το περιβάλλον. Υπάρχουν ε, ανταγωνιστικά προϊόντα, αλλά που δεν είναι ανταγωνιστικά. Μα γιατί μπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καταλαβαίνω. Στην παράγραφο 57 λέει ο κύριος Ζαντό, λυπούμεθα λοιπόν, που το διεθνές εμπόριο ναι. προωθεί προϊόντα που κανονικά θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί τοπικά. Ε, μα ε, ποιος το σκέφτηκε αυτό. Αν ε, είχατε σπουδάσει οικονομία θα γνωρίζατε του κανόνε οικονομία, Η ειδίκευση και το εμπόριο αυτά οδηγούν σε ανάπτυξη ανάπτυξη. Ε, είναι αφελές να σκέφτεστε έτσι και είναι ε, κακό για την παγκόσμια οικονομία οι επιχειρήσεις. Ε, δεν περιμένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δουν τι θα καταφέρει για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Μας επιβάλλει στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν κανένα νόημα από περιβαλλοντική πλευράς. Ενώ η Κίνα και άλλες τέτοιες οικονομίες δεν ασχολούνται καθόλου με το ζήτημα. Και ποιο θα πληρώσει τα σπασμένα με αυτή την ουτοπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εταιρείε και οι πολίτες. Σας ευχαριστούμε, συνάδελφε Στάσεν. Και τώρα θα περάσουμε στους μεμονωμένους ε, ομιλητές ε, από πλευράς ε, των πολιτικών ομάδων, ο κύριος, η κυρία Χάνσλικ. Κυρίες και κύριοι, Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεζιρέ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στα πλαίσια των διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Πιστεύω πως ε, η κοινωνική εταιρική ευθύνη έχει ολένα και ισχυρότερη παρουσία ε, ως προς το διεθνές εμπόριο και το βλέπουμε αυτό από τις πρόσφατες συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Νότιο Κορέα, με την Κολομβία και το Περού χαίρομαι ιδιαιτέρως που το Κοινοβούλιο τονίζει την σημασία του να βασιστούμε σε αυτές τις αρχές για να προστατεύσουμε αυτήν την ιδέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ούτω ώστε να εφαρμόζεται σωστά από τι εταιρείε. Νομίζω ότι αν συμπεριλάβουμε, συμπεριλάβουμε μία ρήτρα στι διεθνεί εμπορικέ ε, συμφωνίε, τελικά ε, θα Έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Θα ενθαρρύνουμε τις εταιρείες να χρησιμοποιούν, να εφαρμόζουν μάλλον ε, με ορθότερο τρόπο τις διατάξεις περί κοινωνικής ε, εταιρικής ευθύνης. Και μην ξεχνάτε ότι οι εταιρείες ε, θα αποφασίσουν αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ή όχι αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο. Ε, οι επιχειρήσεις μπορούν να δεσμευτούν και να υπερβούν κάποιες ελάχιστες δεσμευτικές ρήτρες. Εγώ πήγα στην Ινδία και υπέβαλα αυτή την ερώτηση σε διάφορους επιχειρηματίες επί τόπου. Δηλαδή, ε, τους ρώτησα αν ε, τι προ τίθενται να κάνουν από πλευράς κοινωνικής εταιρικής ευθύνης εκείνη. Μου έδωσαν συγκεκριμένα παραδείγματα γιατί ήδη εφαρμόζουν αρχή της κοινωνικής ευθύνης. Είμαι πάρα πολύ ε, αισιόδοξη και ελπίζω με αυτή την έκθεση του κυρίου Ντεζίρ να ακολουθήσει ένα νέο δρόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να γενικευτούν οι κανόνες, η εφαρμογή, να γενικευτεί η εφαρμογή των κανόνων περί κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε κυρία Χάιντς για τρία λεπτά ο συνάδελφος Κούτας, δεν ξέρω μήπως απαρέφερε το όνομά σας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Ζαντό για την πρότασή του και επίσης για τη διαθεσιμότητά του να συζητά τα ζητήματα με τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι κάποιες στιγμές η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε τη δυνατότητα να μιλήσει με μια φωνή. Η Κοπενχάγη ήταν μια τέτοια στιγμή και όλος ο κόσμος περίμενε να ηγηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει ηγέτης και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει εκείνους που είχαν μείνει πίσω. Όμως ήταν πολύ μεγάλη απογοήτευση. Το συμπέρασμά μα είναι ότι υπάρχει έλλειψη συνένεση εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Υπάρχουν κάποιε κυβερνήσει που δεν είναι έτοιμε να επομισθούν τι ευθύνε του και να αναλάβουν δεσμεύσει για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Μία εξήγηση θα μπορούσε να είναι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που έχει επιβραδύνει ε, την ορμή όλων των φορέων αυτών. Όμω, η καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο και σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να είναι μια συνεχής μέρημνα όλων των κρατών μελών, διότι συζητούμε το μέλλον ε, των επόμενων γενεών. Και μιλάμε και για παγκόσμια δικαιοσύνη. Δεν είναι δίκαιο οι αναπτυσσόμενες χώρες να πληρώσουν το τίμημα της αυξής της δημοκρασίας του και οι βιομηχανικές χώρες να ε, ακολουθούν ρεαλιστική προσέγγιση. Χρειάζεται μια συνοχή μεταξύ Βορρά και Νότου. Η Σύνοδος Κορυφής της Κανκούν ε, αποτελεί μια δυνατότητα για πρόοδο. Θα πρέπει να οδηγήσει σε μια γενική παγκόσμια συμφωνία και νομικά δεσμευτική συμφωνία η οποία θα πρέπει να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας ε, στους δύο βαθμούς ή κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου. Χρειαζόμαστε καλύτερη πολιτική από αυτήν της Κοπενχάγης. Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επίσης δεν μπορούν να εγγυηθούν επιτυχία μετά το 2012. Θα πρέπει να πείσουμε και άλλες χώρες να ακολουθήσουν φιλόδοξες δεσμεύσεις και στόχους. Και τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, ποια είναι η σχέση μεταξύ εμπορίου και αλλαγής του κλίματος. Το εμπόριο είναι πολύ σημαντικό μέσο για την μεταφορά τεχνογνωσίας. Θα πρέπει να εξαλείψουμε τους φραγμούς για το πράσινο εμπόριο. Θα μπορούσαμε να άρουμε δασμού σε επίπεδο ΠΟΕ για πράσινα προϊόντα. Θα πρέπει ταυτόχρονα να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ε, κενό διαφορά μεταξύ των διαφόρων συστημάτων παραγωγής, εργασίας και μεταφορών. Και γι' αυτό θα ενεθάρρυνα τοπική και πράσινη παραγωγή. Ευχαριστώ. Μουτσουμέσκ, αγαπητοί συνάδελφοι Κούτας. Η κυρία Μπέαρμπερ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, η συνέπεια της κοινωνική, της των εταιριών ε, έχει διαδοθεί στον επιχειρηματικό τομέα τελευταία δεκαετία. Πώς μπορεί να έχει αντίρρηση όσον αφορά αυτές τις πολύ βασικές αξίες οι εταιρείε που αντιμετωπίζουν εργαζομένους τους καλά και που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον μέχρι τώρα η σχέση μεταξύ του εμπορίου και της εταιρική ευθύνη, της κοινωνικής ευθύνης των εταιριών ε, δεν είχε ανακαλυφθεί τόσο. Λοιπόν, το διεθνέ εμπόριο ε, είναι στα πλαίσια συμφωνιών μεταξύ κρατών. Εάν θα πρέπει το CSR να είναι δεσμευτική υποχρέωση και θα πρέπει να την υποσυπογράφουν οι εταιρείε ή πρέπει να συμμορφώνονται μόνο εθελοντικά. Οι Ευρωπαίοι πολίτε όλο και περισσότερο καταλαβαίνουν τι γίνεται, ευαισθητοποιούνται. Πρόσφατε είχαμε καταστροφέ όπω και η πετρελοκυρίδα τη BP και έδειξαν υπό ποια, υπό ε, ποια πρότυπα και δοντολογία κινούνται οι ευρωπαϊκές εταιρείες στο εξωτερικό. Πρέπει να ελέγχονται. Και δεν θέλουμε επέκταση στο διεθνές εμπόριο μόνο επί οικονομικών βάσεων όταν το εμπόριο καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και μειώνει το επίπεδο διαβίωσης των τοπικών πληθυσμών. Λέμε ότι φτάνει πια αρκετά. Όταν το εμπόριο καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και μειώνει τα επίπεδα διαβίωσης των τόπιων πληθυσμών, Μόνο οι κυβερνήσει που θα θέσουν προδιαγραφέ που εξασφαλίζουν ότι εκείνοι που συμπεριφέρονται με δοντολογικό σωστά και διαφανή τρόπο δεν βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από εκείνου που δεν ακολουθούν τι προδιαγραφέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει τι επιχειρήσει να υιοθετήσουν και να ενημερώνουν ποιε είναι οι υποχρεώσει για τα CSR σε όλε τι δραστηριότητε επιχειρηματικέ και στη χώρα του και στο εξωτερικό. Και ούτω τρόπο οι κίνδυνοι του CSR, εάν δεν γίνει αυτό, τα CSR δεν θα είναι τίποτα παραπάνω από άσκηση επιχάρτου για δημόσιες σχέσεις, για κάποιες πολυεθνικές. Καλωσορίζω την έκθεση ιδία πρωτοβουλία που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το CSR να το θέσει στο επίκεντρο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι θα σεβαστούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα δικαιώματα των εργαζομένων και ότι αυτά είναι εξίσου σημαντικά επιδιώκοντα τα συμφέροντα τα εμπορικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξωτερικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπέρμπερ. Για ένα λεπτό ο κύριος Ενά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Επιτροπή επειρασπίζεται το άγριο ελεύθερο εμπόριο και έτσι τη διαδραμάτισε το ρόλο της ως επιθύνη οργάνου ε, με δράσεις ε, που βλάπτουν τους πολίτες της Ένωσης. Όντως, εάν ο ανταγωνισμός είναι ελεύθερος, ε, λοιπόν όλα τα ντάμπινγκ είναι εφικτά. Τα φορολογικά, κοινωνικά, νομισματικά περιβαλλοντικά και άρα αναγκαστικά στρεβλώνεται ο ανταγωνισμό. Πώ θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο γιατί ε, οι μισθωτοί και οι οικογένειε τη βυθίζονται στη μιζέρια και ε, όλη η βιομηχανική κλάδη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Τι πρέπει να κάνουν, να καταστρέψουμε του φορολογικού παραδείσους ε, και ε, την ενέργεια, το νερό, τα φάρμακα, τη γεωργία, ε, την ενημέρωση, να τι κάνουμε δημόσιε υπηρεσίε και επίση να τηρούνται τα περιβαλλοντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, ώστε να υπάρχει ισοτιμία ε, στι εμπορικέ συνδιαλλαγέ και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των μισθωτών. Σα ευχαριστούμε, κύριε Νά. Ε, η κυρία Κέστιγκερ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στι τωρινέ αλλά και στι μελλοντικέ εμπορικέ σχέσει έχει μια μεγάλη ευθύνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντο και τα κοινωνικά πρότυπα. Όλα αυτά είναι ακριβώ και βασικά στοιχεία των διαπραγματεύσεων για συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου. Θα πρέπει να τεθούν λοιπόν περιορισμοί και πρότυπα για να εξασφαλίσουμε μια αηφόρο ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν ε, θα θέλω να το τονίσω στον τομέα των σχέσεών μας με την Κίνα και με την Ινδία. Πρέπει να τονίσουμε τα προβλήματα που προέρχονται από την καταστροφή του περιβάλλοντος και από την παιδική εργασία. Θα πρέπει ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε συμφωνίες οι οποίες θα οδηγήσουν σε καλύτερες συνθήκες και πιο πολύ εισόδημα στις χώρες αυτές, αντί να έχουμε απλώς εκμετάλλευση των χωρών αυτών. Αυτά λοιπόν πρέπει να ενσωματωθούν στις συμφωνίες που συνάπτουμε σε εμπορικό πλαίσιο. Δεν πρόκειται μονάχα για ηθικέ αξίε, τι οποίε υποστηρίζει και από τι οποίε εμφορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκειται και για ισότιμη αντιμετώπιση των παραγωγών και μέσα και έξω από την Ευρώπη. Σημαίνει σεβασμό στον Ευρωπαίο καταναλωτή, ο οποίο πρέπει να έχει προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί κάτω από συνθήκε οι οποίε είναι φιλικέ προ το περιβάλλον και ανθρώπινε. Και θα ήθελα να σταθώ και στην έκθεση του κυρίου Ζαντό. Το άρθρο 48 επικρίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο γεωργική πολιτική το οποίο όμως έχει σημαντικό ρόλο για την ποιότητα των τροφίμων. Αναφέρει θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με βλάβες στο περιβάλλον. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων των 500 εκατομμύριων Ευρωπαίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να εξαρτάται από εισαγωγές, πρέπει να έχει μια αυτάρκεια στον τομέα αυτό. Και δεν μπορεί κανείς λοιπόν να ξεχάσει αυτή τη βασική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <coughs> Σας ευχαριστώ. Κυρία Κιώστιγκερ, μπαίνουμε στην οφθαλμοθερευτική διαδικασία. Η κυρία Ρόιτοβα έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με ικανοποιεί η νομοθεσία για το διεθνέ εμπόριο. Θυμάμαι στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή ΙΝΤΕ, εγώ ζητούσε η εμπορική πολιτική να χρησιμοποιηθεί ω ένα εργαλείο για να προωθεί ο θεμητό ανταγωνισμό ε, για την κατοχήρωση των βασικών αξιών και για να προγράμουν τη Ένωση στο διεθνέ εμπόριο. Θέλουμε να ισχύουν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού στον διεθνή ανταγωνισμό. Εδώ πάνω από έξι χρόνια ζητάω όλε οι εμπορικέ συμφωνίε να περιέχουν ρήτρε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ε, ε, ε, ανέκαθεν μιλούσα για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Επιτέλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για την κατάργηση τη εισαγωγή προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προϊόντων που έχουν παραχθεί με παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παιδική εργασία, και αυτό ισχύει για την Ινδία, την Κίνα και άλλες χώρες. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Σάφη. Ε, βλέπουμε ότι σημειώνεται πρόοδος. Καταδεικνύεται αυτό μέσα στην εκθέση. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρόιτεβα. Ο συνάδελφος Νικολάσκη. Σας Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε μετά από την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας έχουμε τη δυνατότητα να πράξουμε πάρα πολλά στον τομέα αυτό, τον εμπορικό και αν θέλουμε να είμαστε ακέραιοι και αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με πιο ενεργό τρόπο συνθήκη συνθήκες Λισαβόνας για να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σημαντικό και από την πλευρά της Κομισιόν <clears throat> να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα έχουν και τις απαραίτητες ρήτρες προστασίας του περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτές οι ρήτρες επίσης θα πρέπει να επαληθεύονται και να εφαρμόζονται με τρόπο αποτελεσματικό. Πρόκειται επίσης και για την προστασία της υγείας η οποία συνδέεται και με την προστασία των ζώντων όντων και θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα την κυρία ε, Σάιφη για την έκθεσή της. Νομίζω ότι μπορούμε να συνοψίσουμε αυτές τις ε, τρεις εκθέσεις λέγοντας ότι χρησιμοποιούνται οι άνθρωποι ε, σαν εργαλείο στις εμπορικές συναλλαγές ε, και παρατηρούμε ότι υπάρχουν μεγάλες απώλειες ως προς το περιβάλλον και ως προς τις οικονομικές ζημιές. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Η ΣΑΕΦ, παραδείγματος χάρη, κάνει καταπληκτικές προτάσεις προτείνει αυξημένο ρόλο για το Διεθνή Οργανισμό Εργασία, ε, καθεστώ παρατηρητού στο ΠΟΕ, μιλάει για τι εκπομπέ αερίων, ε, για διαβούλευση ε, με την κοινή γνώμη. Επίτροπε, αυτά δεν είναι μόνο καλέ προθέσει. Εμεί ζητάμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θέλουμε να πληρούνται οι απαιτήσει μα, θέλουμε να γίνουν οι αλλαγέ που ζητούμε, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τι πρωτοβουλίε ε, Στι ε, διεθνεί εμπορικέ ε, διαπραγματεύσει ώστε να σημειωθεί πραγματική πρόοδο. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Σλίτερ. Και τώρα ακολουθεί ο κύριο Σεγγεντή. Το Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, το κόμμα μου, το UBIC, ανησυχεί τα μάλα και ανησυχεί, ανησυχεί όσον αφορά το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο οικονομική κρίση αυτή που περνάμε, αλλά και περιβαλλοντική και οικολογική που περνάει η Ευρώπη. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι υψής της σημασίας να βελτιώσουμε την κατάσταση και να δούμε τι κάνουν αγωγές αγωγέ ε, τροφίμων. Γιατί χρειαζόμαστε κοτόπουλα από την Βραζιλία και πάπρικα από την Κίνα όταν μπορούμε να τα παράγουμε όλα αυτά στην Ευρώπη. Γιατί χρειαζόμαστε τοπική παραγωγή. Χρειαζόμαστε ντόπια προϊόντα τρόφιμα. Πρέπει να προστατεύσουμε τη βιομηχανία της Ευρώπης, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να προστατεύσουμε τους, πελά, τους πολίτες, συγγνώμη, να εξασφαλίζουμε ασφαλή εφοδιασμό σε τρόφιμα ε, από ευρωπαϊκές πηγές. Πράσινες τεχνολογίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι Σέγγεντη. Τελειώσαμε τη διαδικασία αυτή με τον κύριο Κέλλη του Catch ο κ. Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα, χρειαζόμαστε τον ανταγωνισμό, αλλά πρέπει να ανταγωνιζόμαστε, να υπάρχει σωστό συναγωνισμό. Και κάποιε διευθυντέ που έχουμε τρει χώρε φέρνουν σε μειονεκτική θέση του παραγωγού μα. Η Ελιζάβεθ αναφέθηκε στο Μερκοσούρ. Και πράγματι, πολλά γεωργικά προϊόντα, ηχθείε, αλλιευτικά προϊόντα έρχονται στην Ευρώπη και παράγονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που απαιτούμε εντό τη Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Τούτου λεχθέντο. Κάτι θετικό. Κάποιε από τι συμφωνίε που έχουμε συνάψει πρόσφατα είναι πολύ καλέ. Όπω με την Κορέα. Χρειαζόμαστε περισσότερε τέτοιε. Και συμφωνούν περισσότεροι ότι θα ήταν υποφελέ και για μα και για εκείνου. Τι λέει ο Επίτροπο, θα υπάρξει συμφωνία με την Ιαπωνία οικονομική συνεργασία η οικονομική μελέτη τη Κοπεχάγη έδειξε ότι θα κερδίζαμε 33 δι και εκείνη 18 δι από μια τέτοια ρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Κύριε Κέλλη, συνελήθησαν όλοι οι οφθαλμοί και μπορώ να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Ντεχούχτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. πλουσιότατη συζήτηση. Η φιλοσοφία που διέπει στις εκθέσεις είναι παρόμοια. Οι λεπτομέρειες, οι ιδέες και οι απαντήσεις και οι αποκρίσεις που είδαμε δεν μπορούν να σχολιαστούν ή να απαντηθούν από μένα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλες ιδέες είναι εφικτές, άλλες λιγότερο. Διότι έχουμε και νομικό και θεσμικό πλαίσιο και πολιτικό τέτοιο. Και σαν Ένωση 27 κρατών μελών και σαν μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θα προσπαθήσω να τονίσω τις βασικές πτυχές κάθε εκθέσεως. Δυστυχώς δεν θα είμαι εξαρτητικός. Όσον αφορά την έκθεση Σαΐφη, αρκετοί αναφέρθηκαν στη δυνατότητα θέσεως παρατηρητού του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στον ΠΟΕ. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να βελτιωθούν πολύ και ο συντονισμό και η διεθνή διακυβέρνηση και ο συντονισμό μεταξύ των διεθνών φορέων. Και για να πετύχουμε καλύτερε συνθήκε και αποτελέσματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά μέσω των εμπορικών συμφωνιών χρειαζόμαστε εφικτού στόχου. Οι διαθωτικέ αλλαγέ χρειάζονται χρόνο να εφαρμοστούν. Και αν είναι κανεί ρεαλιστικό όσον αφορά τη συμμετοχή στον ΠΟΕ, αυτό είναι μακρινό στόχο για να συμμετάσχει στο γραφείο εργασία των ε, ΠΟΕ. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση ΣΑΙΦΗ, να γίνονται αξιολογήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπάρχουν σχετικέ εκθέσει στα πλαίσια των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και εγώ θα δίσταζα κατά πόσο μπορούμε να έχουμε ειδικέ περιόδους μεταξύ τέλους των διαπραγματεύσεων και ενάρξεως ισχύω των συμφωνιών. Το συζητήσαμε αυτό και σε άλλο πλαίσιο. Η συνθήκη της Αβώνας καθιστά σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει πρώτα και μετά ξεκινά η διαδικασία επικύρωση που υπογράφει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να επικυρώσει μέσω ψηφοφορίας. Αν πριν τη μονογραφή, πριν την υπογραφή τεθούν κάποιοι όροι, δεν ξέρω, δεν είμαι θετικός. Το να αξιολογηθούν οι συνέπειες μιας συμφωνίας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό έχει κάποια λογική και μπορώ να συμφωνήσω. Ε, τέσσερα συγκεκριμένα ερωτήματα για την εργασία των παιδιών. Διαπραγματευόμαστε τώρα Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με Ινδία. Και πρέπει να τεθεί το θέμα της βιωσιμότητας. Διστάζει πολύ η Ινδία όσον αφορά το κεφάλαιο βιωσιμότητας σε συμφωνίες. Εμείς επιμένουμε όμως και θα συνεχίσουμε. Θέλουμε ένα τέτοιο κεφάλαιο να συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία. Και πιστεύω ότι έτσι θα γίνει τελικά. Αργότερα θα πρέπει να συζητήσετε το θέμα. Παρακαλώ, λάβετε υπόψη. Τι απόψεις έχουν και διάφορες τρίτες χώρες για το κεφάλαιο της βιωσιμότητας. Όχι μόνο όσον αφορά το περιεχόμενο, αλλά και τη φιλοσοφία που ακολουθούν κάποιες τρίτες χώρες. Έκθεση Ζαντού. Άκουσα εκκλήσεις για, κάθε, για κεφάλαιο περικλήματος σε κάθε διμερή συμφωνία. Είμαι υπέρ βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, διότι το μέλλον δεν μας ανήκει. Τι πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να συμπεριφθούν πολλοί παράγοντε για να δοθεί ικανοποιητική απάντηση στην αλλαγή του κλίματο. Χρηματοδότηση, σύλληψη εκπομπών και αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν όμω μέσω διατάξεων σε εμπορικέ συμφωνίε. Υπάρχει ένα ευρύτερο φόρουμ για κάτι τέτοιο. Και αν υπάρχει συμφωνία στο ευρύτερο πλαίσιο, τότε αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στη διμερή συμφωνία για ελεύθερο εμπόριο. Και στον αναπτυξιακό γύρο συζητήσεων, στο γύρο Ντόχα, αν μπορεί αυτά να συμπεριληφθεί, αυτό είναι πιο αμφισβητήσιμο. Διότι δεν συμφωνούν όλοι οι συμμετέχοντε. Σε τέτοιε πολυμερεί συμφωνίε να υπάρχει κεφάλαιο για το κλίμα. Εμείς όμως το υποστηρίζουμε. Τέλος. Έκθεση Ντεζίρ. Πολύ επίκαιρη έκθεση. Διότι είναι ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική ευθύνη των εταιριών είναι κάτι που έχει δρομολογηθεί και ετοιμάζεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέλη του ΟΣΑ συμβάλλουν ενεργά στην ενημέρωση των διαφόρων συστημάτων βαθμολόγησης του ΟΣΑ εν ώψη της διπουργικής του ΟΣΑ τον επόμενο Μάιο. Σε όσες δραστηριότητε σχετικές με τα CSR θα εξετάσουμε προσεκτικά τι διάφορε δυνατότητε προώθηση υπεύθυνης συμπεριφορά των ευρωπαϊκών εταιριών, ανεξάρτητα από το που εδρεύουν και που λειτουργούν, κυρίως όσον αφορά την εφικτότητα και τις συνέπειες και τις ευθύνες. Δεν είναι μόνο εμπορικό ζήτημα, δεν είναι μόνο θέμα διμερών και πολυμερών εμπορικών συμφωνιών. Υιοθετήθηκε πρόσφατα στη ΣΥΠΑ νομοθεσία. Σύμφωνα με αυτή, οι πολυεθνικές με νομική έδρα στην, ε, στη ΣΥΠΑ και όχι μόνο δραστηριότητα στη ΣΥΠΑ θα πρέπει να έχουν ευθύνες, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να παράγουν να κάνουν τις οικονομικές συναλλαγές τους με σωστό τρόπο και σεβόμενοι και τις πρώτες ύλες, βιώσιμο τρόπο. Είναι πρωτοβουλία πολύ αξιέπαινη που είναι εκτός των διμερών συμφωνιών. Η κατεργασία πρώτων υλών δεν είναι κάτι που καλύπτεται κυρίως από διμερείς συμφωνίες. Είναι οικονομικής και βιομηχανικής φύσης δραστηριότητες των πολυεθνικών. Αν η νομική του έδρα είναι στις Ηνωμένες όμως, οι ΗΠΑ μπορούν να δράσουν και να στραφούν κατά των επιχειρήσεων αυτών αν αυτές δεν συμμορφώνονται. Δεν ξέρω, ίσως θα ήταν καλό να κάνουμε και εμείς το ίδιο όσον αφορά τις ε, ευρωπαϊκές εταιρείες που κινούνται στις τρίτες χώρες. Και αν αυτό το επεκτείνουμε και σε χώρες όπως είναι ο Καναδάς, όπως είναι η Αυστραλία. Εν τη αυτή περιπτώσει θα μπορούσαμε να καλύψουμε την πλειοψηφία των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στον κόσμο. Και αυτό θα ήταν μια σημαντική συμβολή όσον αφορά την ανάπτυξη υποβιώσιμου όρους. Συγχαρητήρια για τις τρεις εκθέσεις. Σίγουρα είμαι πρόθυμος να συνεχίσω τη συζητήση επί των θεμάτων τους επόμενους μήνες και χρόνια. Να συζητά μαζί σας δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για να κλείσουμε τη συζήτηση έχουν το λόγο και πάλι δύο λεπτά ο κάθε εισηγητής. Καταρχήν κυρία Σαϊφή έχει το λόγο. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε, Επίτροπε, χρόνο επαρκή στη διάθεσή μας για να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση μετά από αυτά που μας είπατε, οπότε θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, όπως σωστά είπατε, κάποια άλλη φορά. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, ευχαριστώ τους κοιόδους εισηγητές, ευχαριστώ τους συναδέλφους για το και για τη συνεργασία που είχαμε. Ε, ήταν ε, ε, συμπληρωματικά και αλληλένδετα τα ζητήματα και αυτό μας επέτρεψε να συνεργαστούμε και να δούμε τα πράγματα από την ίδια οπτική γωνία. Ε, δηλαδή να εισαγάγουμε την, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα ε, και το περιβαλλοντικό δίκαιο ε, κάπως περισσότερο μέσα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αλλάξουν οι νοοτροπίες, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε να γίνει αυτό από μόνο του. Οπότε, εάν όπως προτείνουμε στις εκθέσεις αγάγουμε σχετικές ερήτρες μέσα στις συμφωνίες, ε, σταδιακά, σιγά σιγά θα διηγηθούμε προς μια πιο δίκαιη, πιο πράσινη ε, οικονομία και θα πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους εμπορικούς της εταίρους. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κυρία Σάιφη. Κυρία Ζαντό τώρα. Και ο κύριος Ζαντό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε Ντεχούχτ για την απάντησή σας και για τις προτάσεις που διατυπώσατε στον τομέα της εργασίας. Εγώ έχω καταγράψει την απάντησή σας για το κλιματικό κεφάλαιο και ελπίζω και για τα άλλα σημεία θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συνεργασία και στη διατύπωση προτάσεων που θα υλοποιηθούν σε συγκεκριμένο επίπεδο στις εμπορικές συμφωνίες μας, διότι σε τελική ανάλυση το γεγονός ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ που είναι πάρα πολύ σημαντικές ότι δεν ευδοκιμούν ναι, αυτό δίνει μεγάλη ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενσωματώσει τις διμερείς συμφωνίες πιο καινοτόμε ρήτρε και πρόνοιες σε ένα νέο τρόπο σύναψη συμφωνιών μια νέα αντιμετώπιση για το κλίμα, για το περιβάλλον, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα κοινωνικά δικαιώματα. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν και υπάρχει μια προσδοκία πολύ ισχυρή προς την κατεύθυνση αυτή. Αν εγκριθούν λοιπόν αυτές οι τρεις εκθέσεις αύριο, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα εξόχω σημαντικό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Απαντώνει στην κυρία Στάσεν για την οικονομία τα εγχειρίδια της οικονομίας εξακολουθούν να γράφονται και τα διακυβευόμενα για το πώς μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα του περιβάλλοντος στο κόστος της παραγωγής, αυτό εξακολουθεί να είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ένα στοιχείο του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Κυρία Κριστίνα, εσείς είσαστε, είμαι μαζί σας όταν υποστηρίζετε την τροφιμική ασφάλεια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά υπάρχουν προσκόμματα με τις συμφωνίες του, του συμφωνίες των ΠΟΕ που εμποδίζουν αυτή την τροφομική ε, επάρκεια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Επίτροπο για όλες αυτές τις προσπάθειες που έχει καταβάλει. Σας ευχαριστώ για να κλείσουμε τη συζήτηση και ο κύριος Δεζίρ. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή είχατε πρόβλημα χρόνου, μπορείτε να μου περικόψετε κάποια δευτερόλεπτα. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Απλώ θα ευχαριστώ του συναδέλφου και να ευχαριστώ και τον Ευρωπαϊκό Επιτρόπο για την απάντησή του. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση είναι η συνένεση που υπάρχει παρά τι διαφορέ απόψεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Παραμένουμε κάποιε αποχρώσει οι οποίε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στι συμφωνίε εμπορικέ, η κοινωνική διάσταση, η διάσταση του περιβάλλοντο. Όταν με είχατε διακόψει, μια παρέμβαση που θα μπορούσε να συναρπάσει ίσως τους ε, συμπολίτες μας. Ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο που ανέφερε και ο κύριος Επίτροπος ότι προφανώς η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει το πνεύμα των νόμων και την ευθύνη των κρατών μελών. Έχει δίκιο βέβαια ο κύριος Δεχούχτ ότι αυτή τη στιγμή και στον ΟΗΕ η έκθεση Ρούτζι που αναφέρθηκε προηγουμένως δίνουν νέες οθήσεις <clears throat> στις προσπάθειες να καθοριστεί η ευθύνη των πολυεθνικών εταιριών σε ό,τι αφορά την εξορυκτική δραστηριότητα, την ευθύνη που επέχουν λόγω των θεατρικών τους στο εξωτερικό και επομένως σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφοδοσίας που εξασφαλίζει τη λειτουργία <clears throat> μιας επιχείρησης και σίγουρα δεν πρέπει να εκφεύγει της ευθύνης μια εταιρεία χρησιμοποιώντας υπεργολαβικές εταιρείε, ή θηγατρικές όταν έχει παραβιάσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα. Όλο αυτό, ε, μάλλον αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναγνωρίζω ότι θα είναι δύσκολο να επιτευχθούν όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον γίνεται μια μικρή και άτολμη ακόμα μνήα της ε, εταιρική ευθύνη τη συμφωνία με τι χώρε της Λατινικής Αμερική και με την Νότια Κορέα, και μετά από όλα αυτά και μετά από τη συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει σήμερα με τον κύριο Επίτροπο, θα πρέπει να προχωρήσουμε για να μπορέσει να υπάρξει μια συνεκτικότητα μεταξύ των στόχων μα στην κοινωνική εταιρική